638 ψήφοι. Απόλυτη πλειοψηφία 320. Σας διαβάζω τις ψήφους που πήραν οι διάφοροι υποψήφοι. Κύριος Λάμστορφ, 393 ψήφοι. Λούνατσεκ, 441 ψήφοι. Ο κ. Παδημούλης, 469 ψήφοι. Πάσκου 517 ψήφοι. Τάραντ 261 ψήφοι. Εκλέγονται κύριοι Πάσκου, Παπαδημούλης, Λούνατσεκ και Λάμπτερτ πέτυχαν την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων. Και βάσει του δεύτερου γύρου έχουν εκλεγεί αντιπροέδροι του Κοινοβουλίου και τους συγχαίρω θερμά τους συναδέλφους αυτούς για το επιτευθέν αποτέλεσμα. Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 του κανονισμού Λοιπόν, η σειρά προτεραιότητα των αντιπροέδρων καθορίζεται από τη σειρά σύμφωνα με την οποία αυτοί έχουν εκλεγεί και σε περίπτωση ισοψηφία από την ηλικία. Η συνθεσία του Προεδρείου θα κοινοποιηθεί στους Προέδρους των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, όσον αφορά την εκλογή των κοσμητόρων, προτείνω να καθοριστεί προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιωτήτων στις 16 ώρα 4 το απόγευμα. Πρέπει να κατεθούν υποψηφιότητε στην Γενική Γραμματεία ε, στο R00101, στο γραφείο R00101, το, ανοιχτό χώρο, το open space τη στο Louis Weiss. Ο πρώτος γύρος ψηφοφοριών θα ξεκινήσει στις 16.30 για την εκλογή κοσμήτωρων. Τα πρακτικά της θεσινής συνεδρίασης έχουν διανεμηθεί, υπάρχουν παρατηρήσεις. Καλώς τα πρακτικά θεωρούνται ως εγκεκριμένα. Λοιπόν, στην ημερήσια διάταξη έχουμε τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου του 2016. Πριν δώσω